Dear colleagues. Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε την ε, συνεδρίασή μας. Με το σημείο 2. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Όπως ξέρετε, η ψηφοφορία για την έκθεση για το σύστημα ανταλλαγής εκπομπών έχει αναβληθεί για την έκτακτη συνεδρίασή μας στο Στρασβούργο την 5η, 15 Δεκεμβρίου, από τις 8 ως τις 10 και θα έχουμε αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, η οποία θα μοιραστεί τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου το απόγευμα. Μοιράστηκε μάλλον ήδη από τη Δευτέρα. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, η αναθεωρημένη ημερήσια μπορεί να εγκριθεί χωρί αλλαγέ. Αναγγελίε του Προέδρου. Προθεσμίζει την υποβολή τροπολογιών. Το σχέδιο έκθεση του κυρίου Στά για την συμφωνία ΣΥΤΑ μετά την αναβολή τη ψηφοφορία στην Επιτροπή ΙΝΤΑ, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ε, στα αγγλικά και μόνο έχει οριστεί για την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου το μεσημέρι. Η ψηφοφορία στην ΕΝΒΗ θα λάβει χώρα στι 12 Ιανουαρίου 2017. Ε, το σχέδιο έκθεση τη κυρία Μέλιν για την προστασία των εργαζομένων από του κινδύνου που έχουν να κάνουν με καρκινογενεί ε, ουσίε και ε, ουσίε που αλλοιώνουν τα κύτταρα έχει αναβληθεί για μία, μετά την έγκριση της πρότασης από την Επιτροπή σε ένα δεύτερο σκέλος υποβολής ουσιαστικών τροπολογιών 21 Δεκεμβρίου 2016 και η προθεσμία ορίστηκε στις 9 Ιανουαρίου 2017 το μεσημέρι. Η ψηφοφορία στην ΕΝΒΗ θα γίνει όπως προβλεπόταν. Μεταξύ των εγγράφων της συνεδρίασης θα βρείτε και μια έκθεση για την επίσκεψη στο Johannesburg στην COP17 του Σάιτες και η οποία έλαβε χώρα από τις 23 ε, ως 25 Σεπτεμβρίου. Το χριστουγεννιάτικο κοκτέιλ. Θα οργανώσω ένα μικρό χριστουγεννιάτικο κοκτέιλ, θα πιούμε ένα ποτό στο τέλος της συνεδρίασης, στην αίθουσα αυτή και όλοι οι βουλευτές αλλά και τα μέλη του προσωπικού ε, είναι προσκεκλημένοι. Σήμερα έχουμε διερμηνία σε 21 γλώσσες και οι συνεδρία όπως γνωρίζετε θα μετατοπεί στο διαδίκτυο. Οι συστάσεις των συντονιστών, σημείο 4 στην διάταξη, έχουν κυκλοφορήσει ηλεκτρονικά. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, τις θεωρούμε εγκεκριμένες. Επίσης, σημείο 5, έγκριση πρακτικών της 29ης Σεπτεμβρίου. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, τα πρακτικά ε, έχουν εγκριθεί. Και τώρα ενημέρωση για τις ενεξελίξει διαθεσμικές ε, διαπραγματεύσεις, κυρίως για τον κανονισμό, για τον Ιδράργυρο ε, Πρώτη φάση ολοκληρώθηκε στον τριμερή διάλογο την 3η 6 Δεκεμβρίου στην συνεδρίαση εκείνη και υπάρχουν σοβαρέ διαφωνίε στα βασικά ζητήματα μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου που θα μπορούσαν όμω να απαλληφθούν. Τα περισσότερα ζητήματα τα καλύψαμε στι συζητήσει για τα νέα προϊόντα και τι διαδικασίε, τα κριτήρια οικονομική αξιολόγηση, όλα αυτά εξαλείφθηκαν και η παρέκκληση για τα επανασχεδιασμένα προϊόντα θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση του υδραργύρου. Επίση, το μέγιστο διάστημα αποθήκευση έφτασε τα χρόνια και η αποθήκευση πάνω από την γη θα έχει να κάνει και με το με τη διαδικασία πρόσθετη σταθεροποίηση. Στι μολυσμένε περιοχέ η Επιτροπή θα δώσει τρία χρόνια για να καταγραφεί ένα κατάλογο από τα κράτη-μέλη για τα προϊόντα που έχουν πρόσθετα υδραγύρου, οι ε, παρεκκλήσεις για τις εξαγωγές θα έχουν οριακές ε, τιμές και αξίες για αρκετά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτάσει στο 2020 την προθεσμία για την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη ευθυγράμμιση στις οριακές αξίες στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τον Υδράγυρο και ιδίω για την ουσία ε, ROHS, για την ένωση αυτή. Ε, στις υπάρχουσες διαδικασίες ε, υπάρχει πολύ γραφειοκρατικό άχθος και γι' αυτό θα υπάρξει μια μεγαλύτερη περίοδος μετάβασης που ε, είναι συντομότερη και από την πρόταση του Συμβουλίου. Για τα πρόσθετα των οδοντικών παρεμβάσεων, οι συνομοθέτες με το Συμβούλιο έχουν προβλέψει μια φάση σταδιακής εξάλληψης. Έτσι υπάρχουν σοβαρές διατάξεις για άλλα σοβαρά ζητήματα, ιδίως με την ηλικία με το όριο ηλικίας 15 ετών για τις ευάλωτες ομάδες, το ποσοστό τήρησης 95% για όλους τους διαχωριστές, τις ημερομηνίες συμμόρφωσης, τα εθνικά σχέδια και το 2020 μια ρήτρα αναθεώρησης για τα στόχους καύσης. Η Προεδρία θα ε, προτείνει το κείμενο στο Κορεπέρ, ε, το υποβάλλει τώρα στο Κορεπέρ, η Προεδρία του Συμβουλίου, και η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΜΒΗ θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου στις 12 Ιανουαρίου. Και τώρα να περάσουμε στην ψηφοφορία. Έχουμε να ψηφίσουμε το σχέδιο ψηφίσματος για την παιδιατρική και τα φάρμακά της. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως ψηφίζοντας την τροπολογία 60. Υπέρ κατά Συνεδραστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 66. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 67. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 68. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 69 με προφορική τριπολογία, που έχει ζητήσει, έχουν ζητήσει οι σοσιαλιστές. Είναι κανείς κατά? Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν, όπως τροποποιήθηκε από τους σοσιαλιστές, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Με συγχωρείτε, 70 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 2, υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Με συγχωρείτε. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Εψήφισαν άπαντες τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 80 ε, υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. Τροπολογία 81 υπέρ. Κατά. αποχέ, έλεγχο. Εψήφισαν άπαντε πέρα Απορρίπτεται. Τροπολογία 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα, ψηφίζουμε από κοινού 6 και 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Καταπίπτει. Καλύπτεται 14 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 τώρα. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα, ψηφίζουμε την 47 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Εψήφισαν άπαντε, πέρα. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικώ. Έλεγχο. Μπορούμε να ψηφίσουμε για την 70 ε, παρακαλώ. Για την 70. για την ε, παράγραφο την ε, καινούργια στη σελίδα 2. Το α νέο. Δεν θυμάμαι αν ψηφίσαμε υπέρ ή κατά. Ψηφίσαμε υπέρ. Νομίζω είπατε κατά για την 70. Έχει, όχι, έχει Εντάξει. Την έχουν προτείνει οι σοσιαλιστές. We have a final vote, sorry. Τελική ψηφοφορία έχουμε, με συγχωρείτε λίγο. Ε, αρχίζει η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Ομόφωνα. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνουμε μια μονόλεπτη διακοπή ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε θέλουν να αποχωρήσουν να το κάνουν. Okay, colleagues. Λοιπόν, συνάδελφοι, περνάμε στο 8. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το Συντορισμό των Οικονομικών Πολιτικών. Ετήσια Επισκόπηση για την Ανάπτυξη 2017. Uh, Θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης του συναδέλφου Νούνο Μέλο. Δεν βλέπω βέβαια τον εισηγητή. Θα δώσω όμως το λόγο στην κυρία Γιούζο. Θα μας παρουσιάσει εκείνη τη θέση του εισηγητού μας. Η Πιλάρ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Νούνο Μέλα, ε, μέλο <laughs> χρειάστηκε να φύγει εσπευσμένα. Μου ανέθεσε όμως να παρουσιάσω εγώ την γνωμοδότησή του, κάτι που κάνω ιδιαίτερη χαρά. Η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο μας δίνει μια εξαιρετική ευκαιρία για την εισαγωγή και περιβαλλοντικών και υγειονομικών πολιτικών στο οικονομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο χάρη μια αηφόρου ανάπτυξη. Η πράσινη οικονομία θα πρέπει να θεωρηθεί ο σημαντικό κινητήριο μοχλό τη οικονομική ανάπτυξη για να μειωθεί η εξωτερική εξάρτηση και να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε με ευφυή και βιώσιμο τρόπο τους σπόρους μας και να μειώσουμε την εξάρτησή μας από την εισαγωγή πρώτων υλών. Βέβαια, οι κλιματικές αλλαγές συνιστούν μια τεράστια παγκόσμια πρόκληση. Εξού και η σημασία της πρόσφατης Συμφωνίας των Παρισίων. Θα πρέπει να παροτρύνουμε συμπεριφορές για βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές και θα πρέπει επίσης να τιμωρούμε όσους ρηπαίνουν ε, ή προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον. Με προφύλαξη όμως, προσοχή, ε, προσπίσοντας την οικονομία, ε, φροντίζοντας για την οικονομική ανάπτυξη και δημιουργώντα προποθέσει για καλύτερη ανάπτυξη σε μερικού κλάδου. Ό,τι αφορά τι ε, πολιτικέ υγεία. Ε, σίγουρα η υγεία είναι ε, αξία από μόνη τη και απαραίτητο προαπαιτούμενο τη οικονομική ανάπτυξη. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε στην υγεία, στο υγειονομικό πλαίσιο, κάτι που θα συμβάλλει στην βελτίωση τη δημόσια υγεία και στην ενίσχυση τη κοινωνική συνοχή. Επίση, θα πρέπει να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας μας. Οι πραγματικές επενδύσεις στην υγεία αποτελεί εκ των όνων κάνευ προϋπόθεση για την οικονομική ευμάρεια και την προώθηση της ανάπτυξης. Για να έχουμε βέλτιστα αποτελέσματα και στην ανάπτυξη αλλά και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ε, προσβλέπω στην αγαστή συνεργασία με όλους τους κοιόδης συγητές. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Γιούσο. Θα ακούσουμε τώρα τους κοιόδης συγητές ο κύριος Ντόφολη από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ανακοίνωση της Επιτροπής για τις Οικονομικές Πολιτικές και την Ανάπτυξη για το 2017 επιμένει σωστά στην ανάγκη να ενισχύσουμε την οικονομική ανάκαμψη, επενδύοντας αποφασιστικά στους νέους και γενικότερα στην καταπολέμηση της ανεργίας. Ε, προκειμένου να συμφωνήσουμε όλοι, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ε, η αδυναμία της Ευρώπης να δώσει ευκαιρίες και προοπτικές στους πολίτες της προφανώς θα δώσει περισσότερες λαβές και χώρο στον λαϊκισμό. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια σωστή συζήτηση στο Κοινοβούλιο ώστε με χειροπιαστές προτάσεις και τολμηρότερες να, να απαντήσουμε στις παλιότερες προκλήσεις που, είναι σε, που αυτή τη στιγμή ε, μεταμορφώνουν τη συνολική εικόνα παγκοσμίω και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πρέπει να χαιρετήσουμε τη θετική κίνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έλλειμμα ανεπολογίζεται στο 2% σε σχέση με το 6% όπως λιγόταν, γινόταν πριν από λίγα χρόνια. Για τη σταθεροποίηση επίσης του δημόσιου χρέους, σωστό και αυτό, αλλά τα διαρθρωτικά κονδύλια εδώ και κάποια χρόνια σε συστάσεις ε, ανακράτος ε, εντοπίζονται και ξεχωρίζονται και σε σχέση με το σύμφωνο σταθερότητας. Θα πρέπει λοιπόν να τα δούμε με διαφορετικό ε, βλέμμα όλα αυτά και να λάβουμε αποφασιστικές αποφάσεις στις πολιτικές απασχόλησεις λόγου χάρη στην οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις επιμέρους βλάβες και ζημιές που έχουν ε, προκληθεί από φυσικές καταστροφές και άλλα τέτοια φαινόμενα. Πρέπει να επενδύσουμε ε, και στην κάλυψη της ευάλωτης φύσης του τραπεζικού συστήματος. Και πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι σε διαφορετικές περιπτώσεις κλειδονισμοί του τραπεζικού συστήματος έχουν να κάνουν και με οικονομικές πραγματικότητες που ε, έχουν φτάσει σε τέλμα και δεν μπορούν να καλύψουν τις πιστώσεις που έχουν αναλάβει οι τράπεζες. Πρέπει να βγούμε λοιπόν από τον ε, ενάρετο κύκλο που έχει δημιουργήσει το δόγμα της λιτότητας. Για τις κοινωνικονομικές μας πολιτικές λοιπόν πρέπει να βρούμε περιθώρια ευελιξίας χωρίς διακριτική μεταχείριση. Και θα πρέπει η ε, λογική του 0, ε, να αντικατασταθεί από την λογική της ποιοτική ε, ανάπτυξης των κρατών μελών, ώστε να φέρουν σε ισορροπία τους προπολογισμούς τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει κάποια μικρά ενθαρρυντικά δείγματα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ως προς αυτό έχουμε πολλά να προτείνουμε διότι πρέπει να επενδύσουμε ε, σοβαρά στην πράσινη οικονομία, έναν από τους τομείς της οικονομίας που έχουν ε, πολύ δυναμικό χαρακτήρα και τη δυνατότητα να παράγει οικονομική ανάπτυξη με δυνατότητες δημιουργίας καινοτομίας και ανάπτυξη στο συγκεκριμένο σύστημα της Ένωσης. Η κυκλική οικονομία, η ανακύκλωση των απορριμμάτων, η μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα με χαμηλές εκπομπές είναι επενδύσεις απαραίτητες από περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης και δεν μπορούμε να τις εγκαταλείψουμε. Για να αλλάξει το μοντέλο μας πρέπει να σεβαστούμε τη Συμφωνία των Παρισιών όπως την ενέκρινε η COP22. Υπ' αυτήν την έννοια τις μνήες ε, στο Παρίσι και την ανάγκη βιωσιμότητα και ανάπτυξη που συλλαμβάνονται στην, ανάγκη της, στην ανακοίνωση της Επιτροπής, τις ε, βλέπουμε πολύ θετικό βλέμμα ε, το ίδιο και την προστασία των πόρων. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε ώστε οι περιβαλλοντικοί δείκτε να μην είναι απλώ στα χαρτιά ωραίε εικόνε και σύμβολα, αλλά πραγματικά κριτήρια για την αξιολόγηση της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. ευχαριστούμε κύριε Τζοφόλη. Ο κύριο Σελίμωβιτς τώρα. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Νουνομέλο, για την γνωμοδότησή του που αποτελεί εξαιρετική βάση για περαιτέρω συζήτηση. Ε, χαίρομαι που εκφέρουμε τη γνώμη μας για την ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη, γιατί τα ενδιαφέροντα ζητήματα είναι ένα τμήμα τη λύση ε, για τα τρέχοντα οικονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα. Και σίγουρα με περαιτέρω πρασίνισμα της οικονομίας θα μπορούσαμε να διορθώσουμε τις ζημιέ που προκάλεσε η κρίση στην οικονομία μας. Θα ήθελα να σταθώ σε τρεις τομεί που κατά τη γνώμη μου έχουν μεγάλη σημασία. Καταρχήν, ε, περιβαλλοντική φορολογία και τα συστήματα μεταφοράς ε, φορολογίας αμεταρρύθμιση της ε, περιβαλλοντικής φορολογίας. Αυτό είναι μείζο πολιτικό θέμα και θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, όπως φαίνεται και από τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Η πρόοδος αυτή θα ρίθηκε κυρίως ε, και από την οδηγία του 2003 για την περιβαλλοντική φορολογία και την μεταβατική περίοδο ε, για την εκπνοή στο μέτρο που οι χώρες θα υποχρεωθούν να εφαρμόσουν νέα φορολογία για τα ενεργειακά προϊόντα. Επίσης, ε, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα της αγοράς, όπως ε, παρατεταμένη ευθύνη των παραγωγών, ιδιαίτερα για τη διαχείριση των αποβλήτων. 25 από τα 28 κράτη-μέλη το 2015 χρησιμοποιούσαν φόρους χωματερή στα πλαίσια της πολιτικής τους για τη διαχείριση των αποβλήτων. Βέβαια, πιστεύω ακράδαντα ότι θα μπορούσαμε πολλά περισσότερα να κάνουμε, ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να μεταφέρουμε το, την περιβαλλοντική επιβάρηση από τους εργαζόμενους στους παραγωγούς και στους ρηπαίνοντες. Και με τη φορολογική, περιβαλλοντική φορολογία θα βελτιώσουμε και την κατάσταση του περιβάλλον και θα βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση, την κατανάλωση στην ενέργεια και θα δώσουμε και κίνητρα ε, για την καινοτομία. Επίσης, ε, ο ρόλος ε, των πράσινων θέσεων εργασίας, των φιλοπεριβαλλοντικών θέσεων εργασίας και μια μελέτη του 2012 έχει καταδείξει ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις οικολογικές βιομηχανίες είναι 3,4 εκατομμύρια για το 2012 και το 2000 ε, είχαμε μόνο 2,2 ε, εκατομμύρια. Βλέπετε ότι αυξάνεται ο αριθμός των φιλοπεριβαλλοντικών θέσεων εργασίας ε, και μάλιστα οι περισσότερες από αυτές εξαρτούνται από το περιβάλλον ως βασικό παράγοντα εισρώης. Για Έχουμε και άλλες πολιτικές την οδηγία του 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων που απαιτεί μέχρι το, ε, την 31η Δεκεμβρίου του 2020 όλα τα κτίρια να έχουν ενεργειακή μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. Επίσης, χρειαζόμαστε καλύτερη απομόνωση και αντλίες θέρμανσης η πρόταση που θα σημειώσουμε στον κλάδο αυτό θα εξαρτηθεί άμεσα και θα υποφεληθεί φυσικά από σωστή εφαρμογή των πολιτικών, όπω αναφέρεται και στις ε, μελέτες που σας ανέφερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πράσινε επενδύσει, επενδύσεις, χρειαζόμαστε όλο και περισσότερες επενδύσεις ε, στο περιβάλλον για να προωθήσουμε τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη. Και παρόλο που οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ έτειναν περισσότερο προ τη δημοσιονομική πειθαρχία, κάτι που ήταν απαραίτητο στα πλαίσια τη χρηματοοικονομική κρίση. Θεωρώ ότι οι επενδύσει είναι αυτέ που χρειάζονται για να υλοποιήσουμε την πράσινη οικονομία που επιζητούμε και θέλουμε βασικού παράγοντε ενέργεια, κλίματο και περιβαλλοντικών πολιτικών στο πολιτικό μα μείγμα. Επίση, οι επενδύσει ε, οι φιλοπεριβαλλοντικές πρέπει να φτάσουν στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να συγκρατήσουμε τη θέρμανση του πλανήτη κάτω από τους δύο βαθμούς Κελσίου. Η ΔΕΜΗ θα περάσουμε σε μία μη αντιστρέψιμη διαδικασία καταστροφική για το κλίμα. Ενώ εμείς υστερούμε κατά πολύ σε σχέση με τις απαραίτητες επενδύσεις σε ε, φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες. Θα πρέπει να βρούμε εναλλακτικού τρόπου για να χρηματοδοτήσουμε τη φορολογία τη πράσινη οικονομία και να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των περιβαλλοντικών φόρων και των επενδύσεων που απαιτούνται και οι οποίε θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσοδοφόρε. Θα πρέπει να είναι ελκυστικέ οι επενδύσει στην πράσινη οικονομία και αποδοτικέ. Θα καταθέσω και κάποιε τροπολογίε στη γνωμοδότηση και περιμένω τι συζητήσει με τους και οδησηγητές μετά την κατάθεση των τροπολογιών. Ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή μας για το πολύ αξιόλογο έργο του. Σας ευχαριστούμε. Κύριο Σέικχαουτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και από τη δική μου την πλευρά ευχαριστώ τον εισηγητή που συνέταξε την έκθεσή του. Είναι πολύ σύντομη γιατί είμαστε περιορισμένοι σε αριθμό χαρακτήρων, ξέρω τους κανόνες, αλλά όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι είναι όντως πολύ καλή η βάση αυτή για να συνεχίσουμε τις συζητήσεις, γιατί όντως θεωρώ ότι είναι κρίσιμη σημασία και χαίρομαι που η Επιτροπή Περιβάλλοντος συμμετέχει στο εξάμεινο αυτό, γιατί όντως ε, αυτό ξέρουμε ότι είναι η μεγάλη οικονομική διακυβέρνηση που ουσιαστικά έχουμε στην Ευρώπη και όπου προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι κυβερνήσεις θα κάνουν ε, έξυπνες κινήσεις με τους προϋπολογισμούς τους ε, και σε περιβαλλοντική, από περιβαλλοντική πλευρά και από πλευρά ε, βιωσιμότητας. Αν δούμε τώρα την πρόταση του εισηγητού σε πολλά από τα θέματα, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε και μάλλον ε, κάποια σημεία θα χρειαστούν απλώς κάποια διευκρίνηση. Και ας πούμε που λέει ο συγκεκριτή ότι οι αρχές της ε, ε, κυκλικής οικονομίας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο εξάμεινο. Ναι, βεβαίως, συμφωνούμε, αλλά θα πρέπει αυτό να είναι πιο ξεκάθαρο. Δηλαδή, τι εννοούμε με αυτές τις αρχές. Γιατί ας πούμε στη συζήτηση για το πακέτο για τα απόβλητα συζητούμε για δείκτες. Είναι σημαντικό αυτοί οι δείκτες να αντικατοπτρίζονται και στο εξάμεινο. Οπότε θεωρώ ότι θα γίνουν κάποιε τροπολογίε για να είναι τα, θέματα, τα πράγματα πιο α, συγκεκριμένα. Για την φορολόγηση, όντω είναι σαφέ ότι είναι δύσκολη συζήτηση πάντα, αλλά όπω είπε και ο συνάδελφο, δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε για τη φορολογία. Αυτό που είδαμε να συμβαίνει κατά τη διάρκεια τη κρίση είναι ότι η φορολόγηση τη εργασία έχει αυξηθεί και είναι πραγματικά ανόητο. Είναι το πιο ανόητο που θα μπορούσε να κάνει κανεί. Γιατί πρέπει ουσιαστικά να μειωθεί η φορολογία επί τη εργασία για να υπάρξουν περισσότερε θέσει εργασία. Και μετά πρέπει να περάσει η ε, φορολογήση στην ε, μόλυνση και, στις, και στους πόρους. Όταν μιλούμε για οικονομία ε, με παρκείς πόρους πρέπει να δούμε ποιο είναι το κόστος και αυτό έχει να κάνει πάντα με τους, με τους πόρους. Οπότε το να μεταφέρουμε την, μετα, την φορολόγηση προ αυτού του τομεί είναι σημαντικό. Επίση, για τι επιδοτήσει για τα ορυκτά καύσιμα. Ε, πραγματικά με έχει κουράσει αυτή ότι αυτές οι διεθνείς πλατφόρμες που συμφωνούν διάφοροι να καταργηθούν αυτές οι επιδοτήσεις. Έχω ε, σταματήσει να μετράω πια πόσες φορές έχουμε πει να το κάνουμε αυτό. Η G20, η G8, ο ΩΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα, όλοι το, το IMF, όλοι το λένε και κανείς δεν το κάνει. Νομίζω λοιπόν ότι τώρα είναι η στιγμή να μπει ένας τέτοιος δείκτης επίγοντος χαρακτήρα στο εξάμεινο για να μην μιλάμε μόνο για την κατάργηση των ε, επιδοτήσεων αυτών, αλλά όντω να το κάνουμε. Οπότε πραγματικά προσβλέπω συζήτηση για αυτό. Ε, θα δω τις ε, τροπολογίες των συναδέλφων για τι πράσινε επενδύσει, γιατί νομίζω ότι εκεί μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πολλά. Και κλείνοντα να πω ότι θα υποβάλουμε κάποιε τροπολογίε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ένα ελάχιστο επίπεδο α, ε, υγείας και πρόνοιας στις χώρες. Ξέρουμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Αν δείτε τι συμβαίνει εκεί, πραγματικά τα βασικά στοιχεία πρόνοιας, εξαφανίζονται ουσιαστικά και φτάνουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα του εξαμήνου. θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας της πρόνοιας. Και αν δείτε και την ασφάλεια ε, της ε, τροφοδοσίας, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για, την, για τα κράτη-μέλη. Η Ευρώπη δεν, δεν πρέπει να μιλά μόνο για μειώσεις οικονομικές, αλλά πρέπει να μιλούμε και για ε, ασφάλεια επισκεπτισμού στην Ευρώπη. Θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες που να το εξασφαλίζουν αυτό. Αν δεν ε, μπορέσουμε να διευρύνουμε το σύστημά μας ε, και συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε μόνο στη λιτότητα, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε σωστά το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην έκθεση. Εγώ με χαρά θα συνεργαστώ και με τους συναδέλφους και με τον εισηγητή, γιατί πραγματικά έχει δημιουργήσει μια πολύ καλή βάση. Θα ε, προσθέσουμε κάποια σημεία για να γίνει η έκθεση πιο συγκεκριμένη, αλλά νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια πολύ καλή γνωμοδότηση που θα πάει στους συναδέλφους της ΕΚΟ. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Τορνάνο. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για το έργο του. Αλλά αντίθετα, με το ειδηλιακό το οποίο μας παρουσιάζει η έκθεση, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχει γίνει τα τελευταία χρόνια το βασικό εργαλείο ε, μιας ε, ενός ελέγχου των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών. Αντί για επενδύσεις σε τομείς υγείας ε, ή παιδείας, η πολιτική λιτότητα οδήγησε στην καταβαράθρωση των δημοσίων υπηρεσιών πολλών κρατών μελών με δραματικές κοινωνικές και υγειονομικές συνέπειες, ιδιαίτερα τη Νότια Ευρώπη. Πέραν της ανάπτυξης και της απασχόλησης, καθώς και της οικονομικής ευημερίας που ζητούμε στην έκθεση, το αντίθετο είχαμε τελικά με την πολιτική λιτότητα. Οπότε δύσκολα προσυπογράφουμε αυτή την αρχή και δύσκολα μπορούμε να ασθενιστούμε τις προτάσεις του επί της ουσίας. Τι να πούμε για αυτό το αμάλγαμα των αντιφατικών προτάσεων που είναι αντιφατικές και με άλλες πολιτικές που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυκλική οικονομία καταρχήν, όντως οι δηλητηριώδεις συνέπειες ε, της, του τρόπου ζωής μας ό,τι αφορά την κατασπατάληση των πόρων είναι αμφισβήτητες, αλλά ε, η γνωμοδότηση λέει ότι βραχαία κυκλώματα θα επιτρέψουν στις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν περίπου 600 δισεκατομμύρια το χρόνο. Η ε, ενθάρρυνση της ε, κυκλικής οικονομίας δεν εννοείται όμως ε, με σύσφυξη του κλειού των επιχειρηματιών, κυρίως με τα όρια εκπομπών, ενώ ήδη οι επιχειρηματίες υποβάλλονται στον αθέμητο ανταγωνισμό της φιλελεύθερης εμπορικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και που αποτελεί την βασική προϋπόθεση και αιτία της παγκόσμιας ρήπανσης. Θα πρέπει σίγουρα να προστατεύσουμε την τοπική κλίμακα, προστατεύοντας όμως και απελευθερώνοντας τις καινοτόμες μας δυνάμεις, δηλαδή τους βιομηχάνους και τους παραγωγούς μας. Άλλος ευσεβής πόθος, αυτός της ενεργειακής αυτάρκειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από ό,τι φαίνεται τα ευρωπαϊκά κρατημένη από μόνα τους δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες και τα ε, ορυκτά καύσιμα σίγουρα δεν είναι ε, ατέρμονη λύση και οι πηγές ανανεώσιμες, ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αποτελούν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Σίγουρα έχουμε πρόθεση, έχουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη, αλλά σίγουρα η απεξαρτητοποίηση από τους προμηθευτές είναι ουτοπία. Επίσης, ε, έχουμε σημαντικές οικονομικές προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη, αλλά οι πόροι μας ε, ε, δυστυχώς δεν αρκούν. Και αυτό θα προ... καταθέσουμε και εμείς φυσικά ε, τροπολογίες στη γνωμοδότηση μέλο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανένας άλλος να θέλει το λόγο. Να δώσω το λόγο στην Επιτροπή, στον κύριο Κλάναγκαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησης και τους κοιόδης εισηγητές για τα σχόλια που έκαναν για την, αίτηση, για την έκθεση για το 2017, για την ετήσια ανάπτυξη εκτιμούμε τα σχόλια που έχει κάνει και τα θέματα που έχει θέσει στην εκθεσή του εισηγητή και βεβαίω την στήριξη που υπάρχει για του ε, τομεί που έχουν ε, τονιστεί ω ε, προτεραιότητα στην έκθεση ετήσια ανάπτυξης που είναι οι τρεις πυλώνες του τριγώνου. Η επανεκκίνηση των επενδύσεων, οι διαθετικέ μεταρρυθμίσει και η εξασφάλιση των σοφρόνων δημοσίων οικονομικών. Στην γνωμοδότηση του εισηγητού ε, πρέπει να συμφωνήσουμε και εμείς για τους στρατηγικούς τομείς ε, που είναι όντως η δημιουργία ε, θέσεων εργασία και ανάπτυξης στην νέα αγορά. Κάποιοι ομιλητέ είπαν ότι η πρόοδος θα εξαρτηθεί και από μέτρα που θα ληφθούν από την πλευρά των κρατών μελών για να αντιμετωπίσουν τα αναπομείναντα εμπόδια στις επενδύσεις, οπότε θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να λάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Καλωσορίζουμε την αναφορά που γίνεται στο σχέδιο έκθεσης ε, στην ε, Συμφωνία για την ε, Κλιματική Αλλαγή των Παρισίων. Η συμφωνία αυτή αναφέρεται ρητά στην ανακοίνωση του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ετήσια έκθεση πρόοδου, γιατί πραγματικά δίνει τις δυνατότητες για τις επιχειρήσεις που μπορούν να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, που σημαίνει συμβολή στην επίτευξη των στόχων που έχουν συμφωνηθεί. Τέλος, για το θέμα των επενδύσεων στην υγεία που ανέφεραν κάποιοι ομιλητές και τον αντίκτυπο στην παραγωγικότητα, την, ε, το κεφάλαιο και την ε, αγορά εργασία. Συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι όντω η υγεία και τα συστήματα υγεία είναι τομεί κλειδιά που πρέπει να, με, το με του οποίου πρέπει να ασχοληθεί το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα και τη βιωσιμότητά του και βεβαίως περιμένουμε ότι ο τομέας της υγείας θα συνεχίσει να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και στις επιμέρους αναλύσεις των κρατών μελών και θα υπάρχει βεβαίως και σε όλες τις εκθέσεις ανάπτυξης. Προσβλέπουμε στην ε, τελική ε, εκδοχή της έκθεσης, ε, συμπεριλαμβανομένων και των όποιων τροπολογιών συμπεριληφθούν και βεβαίως θα περιμένουμε την τελική έκθεση που θα αποσταλεί τελικά στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, για το χρονοδιάγραμμα. Ε, τροπολογίες υποβάλλονται μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου στις 12. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΜΒ έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιανουαρίου και η ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ θα πάει για τις 6 Φεβρουαρίου. Τώρα, πάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσιας διάταξης. Οι απαλλαγές ε, του Γενικού Προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τις υπηρεσίες που είναι υπό τον έλεγχό μας και θα δώσω το λόγο αμέσως στον εισηγητή, σε μένα δηλαδή, για να σας εξηγήσω το σχέδιο έκθεσής μου. Και ζητώ συγγνώμη, αλλά θα περάσω στα Ιταλικά. Μια φορά συμβαίνει και αυτό να θυμηθούμε ότι η ελοποίηση και εκτέλεση του προπολογισμού 2015 ή μάλλον η εκτέλεση και απαλλαγή του 2015 βάσει και τη έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και μετά τις επαφές που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους οργανισμούς που συνεργάστηκαν μαζί μας και ε, ανταποκρίθηκαν με τρόπο ικανοποιητικό στα αιτήματα πληροφόρησης που στείλαμε, Μα οδηγεί στα εξή. Να θυμίσω ότι το 2015 ήταν ο δεύτερο χρόνο εκτέλεση υλοποίηση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου του 2014-2020 και κατά επέκταση, κατά συνέπεια μάλλον, υπήρξαν κάποιες περικοπές σε κάποιες δημοσιονομικές γραμμές σε σχέση με προηγούμενα έτα σε, κάποιε σε κάποιες ε, συγκεκριμένες γραμμές σε σχέση με άλλα έτη και σε άλλε περιπτώσει υπήρξαν αύξηση. Φτάσαμε στο επίπεδο εκτέλεση 99,9%. Αυτό θα πει ότι αξιοποιήσαμε πλήρω τα κονδύλια που είχαμε στη διάθεσή μα. Το επίπεδο εκτέλεση ήταν πραγματικά υψηλότατο. Περνάω απευθεία στα επιμέρου στοιχεία ε, εκτέλεση που μα αφορούν. Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις μέσω της Γενικής Διεύθυνσης ε, ε, Περιβάλλοντος 369.251 ε, εκατομμύρια έφτασαν στο επίπεδο εκτέλεσης 99,36% με τι ε, πιστώσει πληρωμών. Αυτέ οι πιστώσει είχαν επίπεδο χρήση 99,36%. Η Γενική Διεύθυνση Κλίμα αύξησε σε 99,72% το επίπεδο απορρόφηση. Σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία, η Γενική Διεύθυνση Σάντε ήταν υπεύθυνη για ένα <clears throat> πολύ υψηλό ποσό 200.000 εκατομμύρια και το πρόγραμμα δημόσιας υγείας του 2014-2020 επίσης είχε επίπεδο εκτέλεσης πολύ υψηλό 99,9% 72%. Και όλα αυτά αξιοποιήθηκαν πλήρω. Σε ό,τι αφορά την επισητιστική ασφάλεια και την ασφάλεια των ζωοτροφών, κατά την άσκηση, την περίοδο αυτή, τα επίπεδα εκτέλεσης ήταν πολύ υψηλά με κάποια επιπλέον στοιχεία που ενίσχυσαν το Ταμείο Κατεπίγουσων Αναγκών. αναγκών. Όλα εκτελέστηκαν πλήρως. Το 2015 δεν εγκρίθηκαν νέα προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις. Μόνο μία προπαρασκευαστική δράση προβλέφθηκε για τη μεταφορά των ζώων και εξοικονομήθηκαν μάλλον ε, μειώθηκαν οι πρωτοβουλίες για τα επόμενα χρόνια. Σε ό,τι αφορά τώρα τους πέντε ε, αποκεντρωμένους οργανισμούς που αφορούν την ε, αρμοδιότητα της Επιτροπής μας, ΕΦΣΑ, ΕΜΑ, ECDC και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, καθώς και τον ΕΤΣΑ, Ο τεχνικός και επιστημονικός τους χαρακτήρας και πάλι συνοδεύτηκε από μια μεγάλη εκτέλεση και καλή υλοποίηση των πολιτικών. Οι ανθρώπινοι και οι δημοσιονομικοί πόροι αξιοποιήθηκαν καταλήλως για να επιδιωχθούν οι σωστοί στόχοι. Ήταν καλύτερη εκτέλεση του προπολογισμού φέτο, εκείνη τη χρονιά του 2015 σε σχέση με αλέτη. Χρειάζονται κάποια διαφορετικά μέτρα βάσει των συστάσεων και του Κοινοβουλίου και του Ελληνικού Συνεδρίου. Κυρίω ω προ τη συνολική αυτοαξιολόγηση τη μεθόδου εσωτερικού ελέγχου και τα πολιετή προγράμματα. Χρειάζονται περισσότερε λεπτομέρειε και για του διαγωνισμού και για τι υπεργολαβίε. Το ίδιο και για την γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου στην ε, διαδικασία της απαλλαγής του 2014 στον τομέα του δημοσιονομικού ελέγχου και με συγκεκριμένη προσοχή στην ΕΦΣΑ οι εμπειρογνώμονες και οι επιστήμονες συνεργάτες πρέπει να προστατεύονται και από τις ε, αρμόδιες αρχές. Θεωρώ λοιπόν ότι βάσει και των στοιχείων που έχουμε μπροστά μας και όσο μας λέει το ελεκτικό συνέδριο, ε, η απαλλαγή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δαπάνες ε, στους τομείς δημόσιας υγείας, κλιματικών αλλαγών, επιζητιστικής ασφάλειας, υγείας των ζώων και των ανθρώπων και περιβαλλοντικής πολιτικής μπορεί να δοθεί και το είδε και στους πέντε οργανισμούς που βρισκόνται υπό τον έλεγχο της Επιτροπής μας. Και τώρα να δώσω το λόγο στους κοιόδους εισηγητές. Να ξεκινήσουμε με τη συναδέλφο Κάντεμπαχ. Yeah, ich darf mich beim Bericht... Να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή ε, το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα αυτό. Οι γνωμοδοτήσεις είναι διεξοδικότατες, δίνουν την, ε, αντικατοπτρίζουν πραγματικά την ε, εικόνα της Επιτροπής για το πώς βιώνουμε εμείς και πώς μελετούμε τις εκθέσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου. Τώρα αυτό που πρέπει να παρατηρήσω είναι ότι επί της αρχής έχουμε τις παρατηρήσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου για τις διάφορες υπηρεσίες αλλά ε, κάποιες έχουν περάσει στη φάση της ε, εφαρμογή, κάποιες έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό, ε, γιατί πολλές φορές γίνονται οι παρατηρήσεις, αλλά αγνοούνται. Δεν νομίζω ότι είναι καλό αυτό ως προς την συνεργασία, οπότε τώρα βλέπουμε ότι η συνεργασία λειτουργεί και νομίζω ότι από τη δική μας την πλευρά ε, δεν, έχουμε να αλλάξουμε πολλά. Υπάρχουν ένα-δυο σημεία τα οποία ίσως από την πλευρά των ε, σοσιαλιστών θα θέλαμε να τονίσουμε ή να υπογραμμίσουμε, αλλά επί της αρχής μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις ε, θέσεις που μας ανέφερε ο συνάδελφος Λαβία. Ευχαριστώ. Thank you Σας ευχαριστούμε κύριε Κάδεμπαχ. Ο κύριος Σας ευχαριστώ. Θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες επί των εκθέσεων απαλλαγής, των γνωμοδοτήσεων μάλλον απαλλαγής, που είναι καλές και μας χαροποιούν οι εξελίξεις ως προς την μείωση του ποσοστού σφάλματος. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κανένα δύο πραγματάκια που θα θέλαμε να τα επισημάνουμε με τις τροπολογίες μας. Αυτό απλώ ήθελα να σα αναγγείλω ότι πρόκειται να καταθέσουμε σχετικέ τροπολογίε. Σας ευχαριστώ, κυρία Ντορνανό. Ευχαριστώ. Δύσκολο να μην συμφωνήσουμε με το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τους ε, οργανισμούς που εξαρτώνται από αυτήν. Αναγνωρίζω μια χρηστή ε, διαχείριση που χαρακτηρίζεται από τη μείωση του ποστού σφάλματος, την καλή εκτέλεση των κονδυλίων και μία ε, ορθολογική ε, αξιοποίηση του προσωπικού. Έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες μείωσης ε, του προσωπικού κατά 5% στους οργανισμούς, όπως είχε απαιτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες με ομοιόμορφο όμως τρόπο. Θα ήθελα να επισημάνω πάντως ότι η αποτελεσματικότητα θα πρέπει να κριθεί και με βάση το λόγο απασχόλησης ε, προϋπολογισμού, που ε, ποικίλει ανάλογα με τον οργανισμό και μάλιστα οι οργανισμοί που εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κανονιστική της αρμοδιότητα ενέχουν πρόβλημα νομιμοποίησης και διαφάνειας. Ε, κάποιο οργανισμό, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εξαρτώνται κυρίως από ιδιωτικά κονδύλια. Ε, εξού και κάποιες πρακτικές των οργανισμών αυτών που δεν μας ικανοποιούν ένα επεισόδιο του 2014 για μια αίτηση άδεια ε, θέση εμπορία στην αγορά που είχε συμπληρωθεί με πολύ συζητήσιμο τρόπο από τον Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Επίση, σύγκρουση συμφερόντων, άλλη κατάφορη απόδειξη τη εξάρτηση ε, για κάποιου οργανισμούς όπω την Ανώτατη Αρχή ασφάλεια των Τροφίμων. Ε, Υποβάλαμε αυτή την παρατήρηση, αλλά απάντηση δεν έχουμε λάβει ικανοποιητική. Ε, θα πρέπει οι οργανισμοί αυτοί να δρούμε διαφάνεια με βάση και τα επιστημονικά πορίσματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη θέση σε εμπορία κάποιων θεραπευτικών αγωγών, όπως κάποια εμβόλια. Ε, και σε ό,τι αφορά την ΕΦΣΑ θα πρέπει να λάβει υπόψη τις συστάσεις μας για, τις, για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πολιτική της δημόσιας υγείας θα πρέπει να έχει κατά νου μόνο το συμφέρον των Ευρωπαίων, ενώ φαίνεται από, το, από την γνωμοδότηση απαλλαγής πόσες πιέσεις έχει ε, υποβάλει η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα έχουμε τεράστιο υγειονομικό κίνδυνο εξαιτία τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, είτε λόγω παθογενειών στι χώρε προέλευση, είτε λόγω του συγχρονισμού και συνοστισμού στα κέντρα φιλοξενία και υποδοχή των προσφύγων. Αυτά και θα καταθέσουμε και εμεί τροπολογίε φυσικά. Ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρω όμως ποιος είναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τη Γενική Διεύθυνση ΕΝΒΙ Κλίμα και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, το 2015-2016 είναι έτη ορόσημα και μεταβατικά. Διότι, διότι είναι τα πρώτα χρόνια υλοποίηση του προγράμματο LIFE βάσει τη νέα νομική βάση και ολοκλήρωση των προγραμμάτων βάσει του LIFE συν με την προηγούμενη νομική βάση. Είμαστε ικανοποιημένοι από την ε, εκτέλεση του 2015. Ως προς την εκτέλεση, όπως έλεγα, ήταν καλή η εκτέλεση του προπολογισμού. Είχαμε σαφή βελτίωση στην εκταμείευση των πληρωμών από τη Γενική Διεύθυνση Κλίμα. Έχουν πάρει το σωστό ρυθμό πλοήγησης. Ιδίως για συμβάσεις και νέες μεθόδους όπως την ε, πρόβλεψη για νέα δικαιώματα για την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Πραγματικά ξεπερνάμε το 95% για το σύνολο των δικτών. Ένα θέμα με ένα, μια εξέλιξη πολύ θετική. Και το 2015 δεν υποφέραμε όπως τα προηγούμενα χρόνια από έλλειψη πιστώσεων πληρωμών. Έτσι μπορέσαμε να χειριστούμε τι πληρωμές χωρίς να χρειαστεί να περάσουμε σε καμία αναστολή. Δεύτερο σημείο, το ένομον και το συστηματικόν της εκτέλεσης. Πολλοί από εσάς εντοπίσατε τη μείωση του ποσοστού σφάλματος. Το ελεκτικό συνέδριο στις διμερείς επαφές που είχαμε μαζί τους ε, εντόπισαν κάποια πράγματα και έκαναν συστάσεις, όμως καμία από αυτές τις συστάσεις τελικά δεν συμπεριλήφθη στην τελική έκθεση που δημοσιεύτηκε. Δηλαδή καμία σύσταση δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία ώστε να παρουσιαστεί δημοσίως και στις διμερεί συστάσεις που μας έγιναν από το ελεκτικό συνέδριο και απαντήσαμε και φροντίσαμε να τις υλοποιήσουμε Αυτό ήταν αποτέλεσμα πολλών διαφορετικών παραγόντων. Πρώτον, αυτό που είχε ζητηθεί από το, ελεκτικό από το ελεγκτικό συνέδριο ήταν η απλούστευση. Η απλούστευση και η διευκρίνηση των ε, κειμένων, ιδίω των ε, συμβάσεων, των κειμένων των συμβάσεων που είχαν ήδη υπογραφεί από το 2007 και μετά η καλύτερη παρακολούθηση της φάσης υλοποίησης των ε, προγραμμάτων. Τα αποτελέσματα της λήψης αυτών των μέτρων τα είδαμε ήδη και τα βλέπετε με τα τωρινά σημερινά αποτελέσματα. Τέλος, μια παρατήρηση, διότι στην έκθεση γίνονται αναφορές στο στα πιλωτικά προγράμματα και τι προπαρασκευαστικέ δράσεις που θα πρέπει να επικεντρώνονται σε τομεί που πραγματικά προσφέρουν κάτι το διαφορετικό, κάτι το επιπλέον. Εδώ λοιπόν ένα παράδειγμα που είχαμε το 2015 ήταν το πιλωτικό πρόγραμμα BEST. Ένα πρόγραμμα που στόχο έχει να διατηρήσει τη βιοπικιλότητα στις υπερπόμδιες ε, περιοχές και διαμερίσματα όπως η Γουιάννα, η Κανάρι νήσι, η Guadalupe, και είδαμε να έχουν πολύ καλά αποτελέσματα τα προγράμματα αυτά, πραγματικά πολύ ικανοποιητικά. Θεωρούμε ότι ήταν επιτυχημένο. Να δώσω το λόγο στον συνάδελφο της Γενικής Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ. Ευχαριστώ πολύ για τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ. Έχουμε το πρόγραμμα Υγεία, ε, Τρόφιμα και Ζωοτροφές και όπως είπατε και εσείς καλωσορίζουμε την εκτέλεση που ήταν πολύ καλή ε, το μόνο σημείο κονδυλίων που έμενα να χρησιμοποιεί τα για τα έσοδα των οργανισμών ήταν αυτό που μπορεί να εκτελέσει η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή μόνο στο έτος νη συν Για τα τρόφιμα και ζωοτροφές έγινε μια μικρή επιστροφή. Αυτό λόγω της βελτίωσης της αιτήσιας υγείας στα κράτη-μέλη. Υπήρξε ανάγκη να γίνουν κάποιες επιστροφές διότι οι ανάγκες των κρατομελών μειώθηκαν καθησυχάζω τον εισηγητή ότι προφανώ όταν μα δίνει σχόλια συστάσει στο ελληνικό συνέδριο σε συγκεκριμένου οργανισμού, βεβαίω η Επιτροπή και τα μέλη τη, τα διοικητικά συμβούλια, βεβαιώνονται ότι οι συστάσει αυτέ ακολουθούνται. Ακολουθούνται από προγράμματα δράση τα οποία ε, υλοποιούνται κιόλα. Ευχαριστούμε πολύ. Εάν δεν υπάρχει άλλος κανείς που να θέλει το λόγο, ας θυμόμαστε το χρονοδιάγραμμα. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 14 Δεκεμβρίου το μεσημέρι και η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει 30-31 Ιανουαρίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή το Μάρτιο. Και τώρα θα περιμένουμε ένα δίλεπτο να έρθει η συγγήτρια για το επόμενο σημείο, η κυρία Καμπεθών. Σταματάμε για δύο λεπτά. Και μετά ξανασυγγίζουμε μια άλλη φορά. Συγγνώμη, Πρόεδρε. αυτό το δίλεπτο ε, μπορώ να πω κάτι γιατί δεν είναι στην ε, ημερήσια διάταξή μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ε, τη θέση τη δική μας, της Επιτροπής μας, αλλά και άλλων μελετών, την έχει ε, προσυπογράψει για την σχετική οδηγία και νομίζω ότι αυτό αποτελεί καλή προστασία ευρωπαϊκή έτσι ώστε να μην χρειαστεί να, κάνουμε, να αλλάξουμε κάτι από το refit και να μπορούμε κατευθείαν να περάσουμε στην εφαρμογή. Νομίζω ότι αυτό είναι θρίαμβος, πρέπει να το πω. Είναι θρίαμβος της Επιτροπής μας και πραγματικά πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό. Mr. Ο Ναι, ναι. εγώ θέλω να υπάρχει υποστήριξη. Ζητώ συγγνώμη, αλλά αυτά τα μηχανήματα δεν ξέρω και πώς δουλεύουν, καινούργια ναι. είναι. Συμφωνώ λοιπόν για την χλωρίδα και την πανίδα και τα σχετικά κείμενα. Βεβαίως δεν ξέρουμε από εκεί θα προκύψει, αλλά είτε για τους αγρότες ούτε για, τους, είτε για, τους, για ΜΚΟ είναι σημαντικό. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε κατευθυντήρε γραμμέ εφαρμογή πάνω στι οποίε πρέπει να δουλέψουμε. Και νομίζω ότι και η Κομισιόν πρέπει να συνεργαστεί σε αυτό. Ήμουν πριν από λίγε μέρε στην Σουηδία. Θέλαμε να. Κάνουμε μια, να κάνουμε ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο, είπε η Κομισιόν, εντάξει, ας το κάνουμε. Η ε, Σουηδική κυβέρνηση ήρθε πέντε φορές ε, γιατί κάποιος ε, έπαιζε το, έπαιζε το Θεό στην, ε, στις Βρυξέλλες και έπρεπε να αλλάζει κάθε τόσο το σχέδιο. Αλλά πρέπει εδώ να έχουμε συγκεκριμένα επιστημονικά στοιχεία. Δεν μπορούμε οι πολιτικοί ούτε το κοινοβούλιο να παρεμβαίνει. Ε, και λέω πραγματικά στους, στην Κομισιόν, αν συνεχίσετε έτσι θα αρχίσουν να τρέχουν μακριά από την Ευρώπη οι πολίτες. Και το λέω αυτό και προς τον Επίτροπο Γεωργίας. Thank you for your comments. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας. Ε, δεν ήταν χριστουγεννιάτικες ευχές, ε. Ελπίζω να το καταλάβατε. Οπότε, ε, κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι τώρα, ώστε να έρθει η συγγήτρια για το επόμενο σημείο. Okay, we can uh, restart with the next point in our agenda. Να ξεκινήσουμε με το επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης, που είναι ανταλλαγή απόψεων για τις ε, τροπολογίες για την πρόσβαση στα φάρμακα. Έχουμε λάβει 617 τροπολογίες. δύσκολη δουλειά για την εισηγήτρια για να μπορέσει να καταλήξει σε συμβαστικές προτάσεις. Σας δίνω όμως κατευθείαν το λόγο για να μας αναφέρετε την άποψή σας για τις τροπολογίες που λάβετε και, το, και πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δεν φανταζόμουν ότι θα ξεκίνωσα με τόσο νωρί τη συζήτηση. Ήρθα τρέχοντα από άλλη συνεδρίαση. Όπω είπε και ο πρόεδρο, κατατέθηκαν 617 τροπολογίε. Πολύ δουλειά. Πάντω, μέχρι στιγμή η συνεργασία με του κοιόδη ηγητέ είναι εξαιρετική. Και χάρη σε αυτό πιστεύω θα καταλήξουμε στην απαραίτητη συνένεση, τουλάχιστον ευρύτατη συμφωνία όπως απαιτείται από την περίπτωση αυτή. Για δύο, δύο φορές χρειάστηκε να αναβάλουμε ε, την ψηφοφορία. Πάντως ε, έχουν δημιουργηθεί πρόσφορες συνθήκε και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Ο μεγάλο αριθμό ανθρωπολογιών, 617 όπω είπα, δείχνει το ζωηρό ενδιαφέρον που προκαλεί αυτό το θέμα. Δεν είναι τόσο ε, ένδειξη διαφορών. Υπάρχει βέβαια κάποια διάσταση απόψεων αλλά κυρίως οι πολλές τροπολογίες δείχνουν το μεγάλο ενδιαφέρον που προκαλεί αυτό το θέμα. Και χάρη στις θα βελτιωθεί η πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στα φάρμακα. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Ο αρχικός στόχος της έκθεσης πρωτοβουλίας ήταν ε, να εκφράσει την ανησυχία για τις υπέρογες τιμές κάποιων φαρμάκων και την έλλειψη βιωσιμότητας των υγειονομικών συστημάτων στα κράτη-μέλη. Υπάρχει μεγάλη πίεση για τι για τα φάρμακα στα υγειονομικά συστήματα των κρατών Υπάρχουν και άλλα κριτήρια που επηρεάζουν την πρόσβαση στα φάρμακα. Για παράδειγμα, ανάγκη ε, ερευνών σε κάποιους τομείς. Γιατί υπάρχουν τομείς που προκαλούν τι ε, ε, τις ερευνητικές προσπάθειες και άλλοι όχι. Επίσης υπάρχει γραφειοκρατία, κατακαιρματισμός ε, λόγω της ύπαρξης πολλαπλών συστημάτων αδειοδότησης ε, για τα φάρμακα. Η χρηματοπιστωτική κρίση επίσης αύξησε αυτές τις πιέσεις ε, στις υγειονομικέ δαπάνε. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια ανάλυση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν αυτή την πρόσβαση και να δώσουμε μια λύση για να βελτιώσουμε την πρόσβαση στα φάρμακα. Ελήφθη υπόψη Επίση, το γεγονό τη ανάγκη κινήτρων που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των δικαιωμάτων ε, πνευματική ιδιοκτησία ή κάποιων ε, κρατικών ενισχύσεων, ώστε να έχουμε καλύτερη επιστροφή, καλύτερη απόσβεση και αποδοτικότητα των κρατικών επενδύσεων. Επίση, μιλούμε και για τα γενώσιμα φάρμακα. Σημαντικό τμήμα των τροπολογιών ε, αναφέρεται στα γενώσιμα φάρμακα. Εκεί ζητούμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα σε αυτό τον κλάδο, ενώ ταυτόχρονα θα διαφυλάσσουμε με πιο αποτελεσματικά μέτρα την ανταγωνιστικότητα του κλάδου για να βελτιώσουμε τις τιμές, να μειώσουμε τις τιμές και να βελτιώσουμε την πρόσβαση των Ευρωπαίων στα φάρμακα. Πολλές τροπολογίες αφορούν και την ανάγκη μείωση αυτού του κατακαιρματισμού που υπάρχει, της διαφορετικής αξιολόγηση που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα κράτη-μέλη, της προστιθέμενη αξίας και άλλων κριτηρίων. Αυτό είναι προαπαιτούμενο για να καθοριστεί η τιμή και το σύστημα επιστροφής των ε, δαπανών για τα φάρμακα. Χρειάζεται επίση έρευνα σε πολλούς κλάδους που μέχρι στιγμής δεν έχουν προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γι' αυτό και η σχετική τροπολογία στόχο έχει να ενθαρρύνει την έρευνα σε σχετικά παραμελημένους τομείς. Συνέταξα 60 συμβαστικές τροπολογίες, ε, με τις οποίες καλύπτω ένα μεγάλο τμήμα των 617 τροπολογιών και πιστεύω ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των συμβαστικών τροπολογιών ε, θα επιτευχθεί συμφωνία γιατί ήδη οι περισσότερες πολιτικές ομάδες φαίνονται πρόθυμες να υπερψηφίσουν τις συμβαστικές τροπολογίες. Ποια είναι η κατευθυντήρια γραμμή των συμβαστικών τροπολογιών. Ανάγκη μεγαλύτερη συνεργασία και διαφάνεια των κρατών μελών καταρχήν. Επίσης, μιλούμε για την ανάγκη αξιολόγησης ε, μια νομοθετική πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να αξιολογείται καλύτερη προστιθέμενη αξία ε, και η καινοτομία στα νέα φάρμακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε ότι μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να προηγείται αυτή η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας πριν καθοριστεί η τιμή της επιστροφής, το ύψος ε, της επιστροφής. Επίσης θέλουμε να προωθήσουμε την καινοτομία και ταυτόχρονα και την ανταγωνιστικότητα της φαρμακοβιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μειώσουμε τον κατακαιρματισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μιλούμε επίσης ε, για την ανάγκη ε, αναβάθμιση ή ε, λήψη υπόψη αξία πνευματική ιδιοκτησία και να δοθούν κίνητρα ή να, να εξετάζουμε τη χρήση των κινήτρων για την προώθηση της καινοτομία και κατά πόσο τα κίνητρα και οι επενδύσεις συνάδουν με τους στόχους που έχουμε θέσει. Επίσης, μιλούμε για την ανάγκη δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα. Σε περίπτωση δημόσιων επενδύσεων, ε, ζητούμε εγγύηση της Επιστροφή τη αποδοτικότητας των ε, δημόσιων επενδύσεων για την έρευνα. Επίση θα πρέπει να βελτιώσουμε και να διαφυλάξουμε την ανταγωνιστικότητα στην αγορά των γενώσιμων φαρμάκων και εκφράζουμε και μία σημαντική ανησυχία να εξετάσουμε τις αιτίες, ε, τις αιτίες της έλλειψης ε, φαρμάκων και να ενισχύσουμε τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Έχουμε δύο συμβαστικές τροπολογίες που στόχο έχουν τη διασφάλιση της, ε, τη διασφάλιση των συνοπτικών ε, μελετών ή δοκιμών, fast trial, και επίσης ε, ζητούμε καλύτερη αναθεώρηση του κανονισμού για τα ορφανά φάρμακα, τα φάρμακα δηλαδή και τις σπάνιες νόσους. Αυτά είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία του σχεδίου και νομίζω ότι στα πιο σημαντικά από αυτά θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε τώρα με τους Σκιώδη. Ο κύριος Χάινς πρώτος. Ja, vielen Dank, Frau Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Όντως ε, είναι πολύ καλό το κλίμα μέσα στο οποίο δουλεύουμε, οπότε σας επιστρέφω τα καλά λόγια. Ε, όλοι βεβαίως έχουμε, ανησυχούμε για διάφορες ε, ασθένειες, οπότε νομίζω ότι μόνο προς μία κατεύθυνση μπορούμε να πάμε. Ε, στην αρχή ήμουν λίγο σκεπτικός για το ότι την έκθεση. εξακολουθώ να είμαι λίγο σκεπτικός βέβαια, γιατί μιλούμε για περιορισμένη αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έπρεπε να είχα να ακούσω διάφορα σχόλια από ε, συναδέλφους ε, που τελικά ε, με έκαναν να αλλάξω λίγο την άποψή μου, οπότε για κάποια θέματα νομίζω ότι μπορώ να το δεχτώ και η ομάδα μου επίσης. Και νομίζω ότι αυτό είναι ήδη μια επιτυχία. Υπάρχουν διάφορες ανησυχίες για το κόστος των ασθενειών που πρέπει να το λάβουμε φυσικά σοβαρά υπόψη και το οποίο αυξάνεται συνεχώ, ε, το θέμα τη ε, της που συνεχώ ε, αλλάζει, τροποποιείται, πάει μία πάνω, μία κάτω, το καταλαβαίνω βέβαια. ίσως αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μελέτη ενό εισαγγελέα. Στη Γερμανία συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παίζει πάντα τον, το ρόλο του καθορίζοντα τις τιμές. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες ρυθμίσεις και στη δική μου χώρα που δεν ορίζονται μόνο από την βιομηχανία αλλά υπάρχουν πολλά περίπλοκα συστήματα για τον καθορισμό των τιμών. Συμφωνώ απολύτως για τις χώρες Μπενελούξ, για την Αυστρία, που ακούω ότι ε, δημιουργούν έτσι μια ομάδα για να δημιουργήσουν ε, τους κατάλληλους κανόνες έτσι ώστε να μπορούν να αντισταθούν στην ε, βιομηχανία. Νομίζω ότι είναι καλό αυτό. Και έχουν πραγματικά πλήρως την υποστήριξή μου. Και επίσης είμαι γνώμη που έχουμε νέους ε, σοσιαλιστές που δίνουν το μπαλμό στην έκθεση αυτή. Νομίζω είμαστε στη μέση του δρόμου και μπορούμε να προχωρήσουμε προς τον ε, δρόμο που μας δείχνουν. Ε, βεβαίως να μην ξεχνούμε ότι η φαρμακοβιομηχανία ε, έχει κάνει πραγματικά τεράστια δουλειά σε ό,τι αφορά τις καινοτομίες και ε, δεν θέλω να πω πράγματα που έχω ξαναβεί. πριν από 20 χρόνια είχαμε ασθένειες που οδηγούσαν στο θάνατο. Σήμερα τις αντιμετωπίζουμε πολύ πιο απλά. Βεβαίως πρέπει πάντα να κάνουμε σωστές, ε, εμβριθείς μελέτες ε, και σε αυτό εγώ πάντα λέω ναι. Ε, τώρα, για την βοήθεια σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, νομίζω ότι αυτή είναι καλή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Μπορούμε να έχουμε σωστά αποτελέσματα μέσω συνεργειών. Και βεβαίως υπάρχει και αντίστοιχη δραστηριότητα που γίνεται στο θελοντικό επίπεδο και νομίζω ότι στην, σε πρώτη φάση θα πρέπει να δούμε την προσθέμενη αξία επί τη βάση των επιστημονικών μελετών. Νομίζω ότι οι σοσιαλιστές φίλοι μου και οι πράσινοι φίλοι μου θα θίξουν ε, διάφορα θέματα σε ό,τι αφορά και την ηθική. Τους εύχομαι καλή επιτυχία, γιατί τα θέματα της ε, ηθικής εναρμόνισης μεταξύ βορρά, βορείας, Βόρειας Ευρώπης και Νότιας Ευρώπης δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν να το περάσουν. Ε, βεβαίως αυτό είναι θέμα και των χωρών. Οπότε ας αφήσουμε τους επιστήμονες και τα επιστημονικά κριτήρια που υπάρχουν να δουλέψουν, να τα χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να μην κάνουμε διπλή δουλειά. Πνευματική ιδιοκτησία. Ε, εκεί είμαι λίγο διστακτικός. Ε, αυτοί που έχουν ε, ε, επενδύσει πολλά χρήματα για να εκπονήσουν νέα διπλώματα ευρεσιτεχνία θα πρέπει να καταλήξουν τελικά σε αυτά τα ε, διπλώματα. Έχουμε, οι νέοι μας έχουν καλή εκπαίδευση, ε, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν ε, νέοι που καλλιεργούν ε, διάφορες συσκευές που μπορούν ε, να χρησιμοποιήσουν ε, τις συσκευές αυτές για να κάνουν διαλογή από τα σκουπίδια, σιδήρου και άλλων στοιχείων. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα είδη πνευματικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που μπορούν να προωθηθούν. Δεν νομίζω όμω ότι μπορούμε όσο αφορά την πνευματική ιδιοκτησία να ανοίξουμε πολύ του κανόνε. Ε, Βεβαίω υπάρχουν δυνατότητε να επεκταθούν ε, τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Αν α πούμε λήξει ένα δίπλωμα, ε, μπορούμε λιγάκι να το, να το τροποποιήσουμε κάπως για να υπάρξει μια παράταση παρόλο που μπορεί να υπάρχει, που, δεν μπορεί, που μπορεί να μην υπάρχει κλινική ε, χρήση για τους ε, ασθενείς μας. Για τις τιμέ ε, τα είπα, είπα την άποψή μου και να επαναλάβω για τις χώρες Μπενελούξ, την Αυστρία και κάποιες από τις σκανδιναβικές που έχουν εδώ και καιρό ξεκινήσει να ρυθμίζουν τα θέματα αυτά διμερώς. Νομίζω ότι στην ε, φάση που βρισκόμαστε είμαστε, είναι μια καλή προσέγγιση. Για τα γενώσιμα συμφωνώ απολύτω. Υπάρχουν ε, συχνά γενώσιμα στη δική μου τη χώρα, τα υποστηρίζουμε ακριβώ για τα άτομα που μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν τα άλλα φάρμακα. Ε, τα συμβατικά. Οπότε και πάλι ευχαριστώ την ε, ε εισηγήτρια. Ήταν όντω πολλή δουλειά, αλλά έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Οπότε, κύρια εισηγήτρια, συγχαρητήρια και πρέπει να πω ότι με χαρά συνεργαζόμαστε μαζί σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φαρία, ευχαριστώ πρόεδρε. Περνώντας αφορμή από τα λόγια του συναδέλφου που μόλις παρενέβη, θα ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για τη δουλειά τη καθώς και τους συναδέλφους Κιώδης. Θέλω να πω ευθύς εξ αρχή. ότι ο στόχο είναι να καλυφθούν οι ανησυχίε που είχαμε σε όλο το διάστημα τη δουλειά μα. Το συζητήσαμε και στι συνεδριάσει με του και στι τεχνικέ συνεδριάσει. Και παρά το γεγονό ότι σε κάποια ζητήματα τις αποφάσεις για την επιστροφή της αξίας των φαρμάκων που τις λαμβάνουν τα κράτη-μέλη, το κόστος και η αξία επιβαρύνουν τους προπολογισμούς. Και ιδίως αυτό δυσκολεύει την, τον τομέα της καινοτομία στη φαρμακοβιομηχανία. Πρέπει λοιπόν να δούμε τη βιωσιμότητα της κοινωνικής πρόνοιας των κρατών μελών και το επίπεδο ποιότητας που μπορούν να προσφέρουν και τις απαραίτητες επαναστατικές και καινοτόμες κινήσεις που χρειάζονται στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας στα κράτη-μέλη. Είναι σημαντική και η διεθνής ανταγωνιστικότητα και θα πρέπει να υποστηριχθεί. Γι' αυτό καλό θα ήταν να θυμίσουμε ότι η υγεία θα πρέπει να έχει και μία διάσταση οικουμενική, να εξασφαλίζεται σε όλους και όλοι να έχουν εύκολη πρόσβαση. Η πρόνοια η στέρηση πρόσβαση στην πρόνοια για οικονομικούς λόγους, όπως ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι στις συναντήσεις που είχαμε, είναι απαράδεκτη. Και είναι μία ένδειξη ότι αυτό το σενάριο πολλέ φορέ πολλά, συμβαίνει σε πολλά κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μπορεί να συμβάλλει για να εξορροπήσει και πάλι το, την αγορά των φαρμάκων όπω πρέπει, ώστε να υπάρξει καινοτομία από τον κλάδο και θα πρέπει να υπάρχει ε, εξισορρόπηση της πληροφορία, των πληροφοριών που παρέχουν φαρμακοβιομηχανίε στα κράτη-μέλη ώστε από τη μια οι καινοτόμε εταιρείε να στηρίζονται και από την άλλη η γενική σύγκληση για τις βιώσιμες τιμές των φαρμάκων να, εξασφαλιστεί, να σε σχέση πάντοτε και με την τιμή των ε, καινοτόμων φαρμάκων. Οι επιθετικές ενέργειες στην τιμολόγηση των φαρμάκων είναι από τα κεντρικά σημεία. Όταν μιλάμε για βελτίωση της πρόσβασης στα φάρμακα, το περιθώριο για βελτίωση για βελτίωση τη ε, συνεργασία ε, στην επιστημονική και τεχνική ε, έρευνα είναι κάτι που θα μας επέτρεπε να εξοικονομήσουμε και πόρους ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη προσπαθειών ιδίως στις, στους πόρους των κρατών μελών και να εκμεταλλευτούμε πολλαπλασιαστικά την αξία των νέων φαρμάκων που φτάνουν στην αγορά. Επίσης, αναφέρθηκε ότι η πραγματική καινοτομία παράγει κέρδος για την υγεία για όλε τι οικονομίες και τον κλάδο της κοινωνική του πρόνοιας, τη δημόσια υγεία. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην έχουμε και να έχουν εξωφρενικέ τιμέ τα καινοτόμα φάρμακα, διότι σε αυτή την περίπτωση οι ασθενείς πραγματικά τα χρειάζονται, θα μπορούν να τα ε, προμηθευτούν. Πρέπει να υπάρχει και εκεί ένα έλεγχο. Αυτό ήταν, ε, αυτέ ήταν κάποιε από τι μέρημνε που απασχολούσαν την κοινωνική ομάδα, την άλλη επί του θέματο αυτού. Θα πρέπει να δούμε και τι εθνικέ αρχέ, τι αρμόδιε αρχέ για την απόφαση καθορισμού των τιμών και των επιστροφών. Προκειμένου να έχουμε μοντέλα τιμολόγηση που να είναι πιο βιώσιμα, πιο δίκαια και να προσφέρουν και πραγματικό κερδό στον τομέα τη δημόσια υγεία. Να υπάρχει δηλαδή αξία για του ασθενεί. Θα πρέπει να προσέχουμε πώ καθορίζουμε το κόστο των νέων προϊόντων όπω και τον αντίκτυπο στον προπολογισμό των κρατών. Αλλά όπως είπα όλα αυτά έχουν αναφερθεί όχι μόνο εδώ πολλαπλώς αλλά και στις ε, συνεδριάσεις, τις τεχνικές συνεδριώσεις και τις συνεδριάσεις με τους κοιόδης. Επίσης θα πρέπει να έχουμε εύρωστα συστήματα για την ε, ε, διαρκή και την συστηματική συλλογή δεδομένων για τις νέες διαδικασίες και τα φάρμακα, να βλέπουμε το πώς λειτουργούν τα φάρμακα στον τομέα της υγείας και τα συστήματα να είναι διαλογικά, να είναι συγκρίσιμα τα δεδομένα, ώστε να είμαστε βέβαιοι για την αξιοπιστία και την ε, διεξοδικότητα των δεδομένων προκειμένου να διευκολύνουμε την καινοτομία. Το ίδιο και για το απόρριτο, την εμπιστευτικότητα και για τι συμφωνίε των κρατών μελών. Τέλο πάντων, όλα αυτά που είναι ανησυχίε, τι οποίε έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενε συνεδριάσει και τι γνωρίζει η συγκήτρια. Θα προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε τι διαφορετικέ απόψει των διαφορών πολιτικών ομάδων και τέλο πάντων έχει γίνει πολλή δουλειά ήδη. Θα ήθελα να ολοκληρώσω μιλώντας για ένα σημαντικό πολιτικό σημείο, την σύγκληση. Θα πρέπει το μήνυμά μας εδώ να είναι να αποσαφηνίσουμε λίγο τον επιδιωκόμενο στόχο. Τόσο όπως ήδη ξεκινήσαμε να κάνουμε στις συνεδριάσεις συνοδοσκιώδης, αλλά και στις τεχνικές. Τέλος πάντων, νομίζω ότι τα έχουμε πάει καλά ως τώρα. Θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Ριβαζή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδης ηγετές και τους συναδέλφους για την ανταλλαγή απόψεων. Βλέποντας όμως τον τίτλο της έκθεσης που λέει πρόσβαση στα φάρμακα. Το μείζον πρόβλημα είναι η τιμή των φαρμάκων. Για να έχει κανείς πρόσβαση θα πρέπει να είναι ε, προσιτή τιμή του, φάρμακο, του φαρμάκου, να μην είναι απλησίαστα τα φάρμακα και επίσης να μπορούν οι, ε, οι κοινωνικές ασφαλίσεις να επιστρέφουν ε, τις τιμές αυτές, να επιστρέφουν στους ασθενείς τα φάρμακα. για μια εικοσαετία η φαρμακοβιομηχανία είχε μονοπόλιο και μέχρι το 2000 είχε περίπου ένα δισεκατομμύριο κέρδος το χρόνο. Έκτοτε είχαμε μια πόλη της καινοτομίας και θα επανέλθω στο θέμα της καινοτομίας. Τι έκαναν λοιπόν, ε, ε, δημιούργησαν φάρμακα παρόμοια με αυτά που υπήρχαν και όταν έχουμε ένα μόριο που έχει θεραπευτικές ικανότητες, ε, τα εργαστήρια προσδιορίζουν την τιμή του φαρμάκου ε, και μάλιστα υπάρχουν και θύλακες για φάρμακα για σπάνιες νόσους που εκεί και αν είναι απλησίες ε, οι τιμές. Είναι αστρονομικές τελείως. Γι' αυτό και είπα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να δούμε το θέμα τη πρόσβαση. Ε, υπάρχει το θέμα των υποχρεωτικών αδειών. Γιατί δεν βοηθάτε τα κράτη-μέλη, και εκεί μπορεί να παίξετε ρόλο, να χρησιμοποιήσουν τι υποχρεωτικέ άδειε. Δείτε τι γίνεται στην Ινδία, στη Βραζιλία, στην Αλγερία χρησιμοποιήστε τις υποχρεωτικές άδειες για ένα ε, φάρμακο σαν το σουφοσμπιβίρ ε, μπορεί να ε, κοστίσει από 100 μέχρι 2.000 ευρώ. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Και εκεί μπορείτε να βοηθήσετε τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν τις υποχρεωτικές άδειες. Έτσι θα καταλάβουν και τα φαρμακολογικά εργαστήρια ότι δεν μπορούν να συντρίβουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας των κρατών μελών με τις υπέρογες τιμές. Ό,τι αφορά επίσης τη σύνδεση μεταξύ του προσδιορισμού της τιμής και της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, ε, day linkage, η αποσύνδεση. Έχουμε μία ανεξάρτητη ε, ιατρική εφημερίδα περιοδικό που έλεγε τα τελευταία 40 χρόνια μόνο δύο νέα φάρμακα τέθηκαν σε εμπορία για την καταπολέμηση της φυματίωσης. Ενώ θερίζει 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους το χρόνο. Ενώ είχαμε, εκατοντάδε ε, είχαμε εκατοντάδες φάρμακα για τις αλλεργίες, τις ανοιξιάτικες. Οπότε δεν είναι προτεραιότητα των φαρμακοβιομηχανιών η εξυπηρέτηση της δημόσιας υγείας, αλλά το κέρδος. Τι φάρμακο θα, έχει περισσότερο, θα φέρει περισσότερο τζίρο. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια αποσύνδεση μεταξύ της τιμής και της ε, καινοτομίας ε, και έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Επίση, πώ θα, πώς θα ενισχύσουμε την καινοτομία. Καταρχήν, τι σημαίνει καινοτομία. Ή θα έχουμε ένα επίπεδο εφεύρεση, εφευρετικότητα, Αυτό είναι σημαντικό κριτήριο για την κατανόμη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία και αυτό γίνεται σε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνία, σε επίπεδο κρατών μελών. Είναι σημαντικό, είναι και φυσιολογικό για την καινοτομία. Επίση, η προστιθέμενη θεραπευτική αξία του φαρμάκου είναι πολύ σημαντική. Για παράδειγμα, η τεχνολογική εφεύρεση. Οι γιατροί του κόσμου, με τη saint Μόντ, ε, άσκησαν προσφυγή κατά του ε, γραφείου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ε, με τον ισχυρισμό ότι σου φοσμπιβίρ δεν είναι καινοτομό φάρμακο, δεν περιέχει αυτή την αρχή της καινοτομίας και κέρδισε τελικά την προσφυγή. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάζουμε την θεραπευτική προστιθέμενη αξία. Αυτή όμως εξετάζεται στα, κράτη σε επίπεδο κρατών μελών. Θα πρέπει όμω να ληφθεί υπόψη στον προσδιορισμό τη τιμή και στο επίπεδο τη επιστροφή. Ε, μία τεχνολογική εφεύρεση δεν σημαίνει κατά ανάγκη προστιθέμενη θεραπευτική αξία ενό φαρμάκου. Και το αντίστροφο επίση. Οπότε θα πρέπει να γίνει αυτή η διαφοροποίηση στην έκθεση. Καινοτομία δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι το φάρμακο έχει προστιθέμενη θεραπευτική αξία. Πάντω ε, ακολουθεί καλή άγουσα η έκθεση, αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου το γενικό συμφέρον. Θα πρέπει εμείς ε, από μόνοι μας να καινοτομούμε, γιατί αυτή τη στιγμή τα διπλώματα ευρυστεχνίας δεν ε, είναι εχέγγυο ότι θα έχουμε νέα φάρμακα που ανταποκρίνονται στις ε, ανάγκες υγείας του πλανήτη. Ή θέλουμε κάτι άλλο πέραν των διπλωμάτων ευρυστεχνία ή να παρακάπτουμε τα διπλώματα ευρυστεχνία όταν έχουμε μία έκτακτη υγειονομική ανάγκη ή ε, να δούμε και τι γίνεται σε επίπεδο ΠΟΕ. Δεν θα πρέπει να είμαστε εχμάλωτοι των φαρμακοβιομηχανιών ή των φαρμακολογικών εργαστηρίων. Επειδή είμαι και στην ε, ε, αντιπροσωπεία για την Αφρική, Καραϊβική και Ειρηνικό, ε, μας λένε ότι η Ευρώπη έχει χρηματοδοτήσει τις κλινικές μελέτες και δοκιμές και τελικά οι φαρμακοβιομηχανίες έχουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνία και αυτές προσδιορίζουν τις τιμέ των εμβολίων, για παράδειγμα, σε, υπέρογκες, σε υπέρογκα επίπεδα. Είναι σημαντικό και απαραίτητο να πληρώνουμε ε, τις φαρμακοβιομηχανίες, αλλά θα πρέπει να έχουμε και δημόσιες επενδύσεις για την έρευνα σε τομείς που οι φαρμακοβιομηχανίες στα εργαστήρια δεν θέλουν να επενδύσουν. Ευχαριστώ κύριο Πεντητσίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την ε, συγγετρία, εκτός μικροφωνού. Μικρόφωνο. Έσβησε. Να επικεντρωθώ στο θέμα των ε, παιδιατρικών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε παγκοσμίω 130-150 εκατομμύρια άτομα που έχουν πληγεί από την υπατήτητα γάμα και από όλε τι ασθένειε που αφορούν το σηκώτη και έχουν σχέση με την υπατήτηδα, τρίτη γάμα. Ε, αυτά τα στοιχεία είναι σχετικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι στη Βόρεια Ευρώπη κυρίω έχουμε συχνότητα εμφάνιση 0,1 και 1%, στην ε, με κεντρική 0,2 έω 2% και στην ε, Νότια Ευρώπη 2,5 με 3,5%. Με τέτοιους αριθμούς μπροστά μας, ε, με τέτοια σεβαρή παρουσία σε πολλές περιοχές της Ένωσης, μας φαίνεται περίεργο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν καταφέρνει ακόμα να ξεκινήσει ένα πραγματικό πρόγραμμα δράσης για την ε, καταπολέμηση, την αγωγή κατά της πατήτητας γάμα. Ίσως να μην είναι έτσι. Η δική μας πάντως αίσθηση είναι ότι είναι πιο βολικό να παραμένει ασθένεια αθεράπευτη παρά να αντιμετωπίζεται. Και μάλιστα αντί να προλαμβάνεται η ασθένεια, είναι λες και προσπαθούμε να την κάνουμε ακόμη πιο χρόνια με τι τεράστιε δυνατότητε κέρδους που προσφέρει η καταπολέμησή τη. Και η επιτατήδα Γ μπορεί να εκκριζωθεί. Γι' αυτό οι τροπολογίε μα, γιατί θέλουμε την πρόημη διάγνωση, την έγκυρη διάγνωση και την αντιμετώπιση με τα σωστά φάρμακα. Εδώ και 30 χρόνια, το είπε και η Συνάδελφο Ριβαζή, βρίσκεται στην αγορά φάρμακο το οποίο... αντιμετωπίζει και εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό του ιού, αλλά με τεράστιο κόστος. Στην ε, Ιταλία 40 με 30.000 ε, ευρώ αναγωγή και ασθενή, στην Ισπανία 50.000, στη Γερμανία 30.000, 40 στη Γαλλία. Είναι τεράστιες τιμές, αλλά 267 φορές ε, μεγαλύτερη τιμή από το κόστος παραγωγής. 50 ευρώ θα πρέπει να κοστίζει το φάρμακο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν η δυνατότητα πρωτοβουλία τη συναδέλφου Καμπεθών θα πρέπει να είναι λίγο πιο αποφασιστική και πιο ε, καυστική σε αυτά τα σημεία. Και η Επιτροπή μα, η Επιτροπή ΕΝΒΗ, πρέπει να αποστείλει ένα σοβαρό πολιτικό μήνυμα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι μόνο με ένα πρόγραμμα κατά τη υπατήτητα Γ, που, θα, ε, που εδώ λείπει οποιαδήποτε νομική ευρωπαϊκή παρέμβαση, αλλά προστατεύοντα τα δικαιώματα των ασθενών ε, με έναν τρόπο συνολικό. Όχι μόνο με τη χρόνια αγωγή για την αντιμετώπιση των ε, χρόνων παθήσεων, γιατί αυτό εξυπηρετεί μόνο τι μεγάλε φαρμακοβιομηχανίε. Θα πρέπει λοιπόν να ε, αντιμετωπίσουμε τι αδυναμίε του συστήματο με τρόπο αποφασιστικό και τολμηρό. Και να ακούσουμε και αυτά που η Επιτροπή Αναφορών μα έχει πει, γιατί έχει λάβει πολλαπλέ αναφορέ από του Ευρωπαίου πολίτε, ε, των οποίων απορρίπτεται το δικαίωμα πρόσβαση στα κατάλληλα φάρμακα. Ευχαριστούμε ο κύριο Ντόρφμαν τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Και εγώ έχω υποβάλει κάποιες ε, τροπολογίες για την ε, διασυνοριακή πώληση φαρμάκων. Όντως αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα γιατί ε, εκεί στις διάφορες ε, περιοχές ε, που υπάρχουν πολλοί τουρίστες είναι δύσκολο να φτάσει κανείς να έχει πρόσβαση σε φάρμακα με συνταγές άλλων χωρών. Ξέρω ότι βεβαίως το θέμα αυτό είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Υπάρχουν κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτού του είδους τις πωλήσει μεταξύ φαρμακείων ε, τις επιτρέπουν και τις έχουν ρυθμίσει. Άλλοι όπως η Ιταλία δεν το πράττουν, οπότε κάποιος, ε, ένας φαρμακοποιός στην Ιταλία ε, δεν μπορεί ας πούμε να εκτελέσει μια συνταγή από τη Γερμανία ή από κάποια άλλη χώρα. γιατί ο ασθενή έρχεται με μια ξένη προ τον Ιταλό φαρμακοποιό συνταγή. Οπότε ξέρω ότι αυτό το θέμα είναι εθνική αρμοδιότητα, αλλά εν πάση ίσως καλό καλύτερα να, να πιέσουμε λίγο, γιατί ούτω ή άλλω είναι και ένα κομμάτι τη εσωτερική αγορά που μας αφορά. Ευχαριστώ. Thank you very much, Ευχαριστούμε ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Καμπεθών για την τεράστια δουλειά τη πολύτιμη η ε, προεργασία της και κατέγραψε πολλές από τις δικές μας παρατηρήσεις όλων των πολιτικών δυνάμεων. Την ευχαριστώ λοιπόν για τη δράση της. Κατέληξε σε ένα σοβαρό αποτελέσμα για ένα θέμα Αυτό της πρόσβασης στα φάρμακα. Θεωρώ ότι είναι ένα ντοσχέ θεμελιώδους δημοσίας σημασίας. Διότι η οικονομική κρίση, κατά την άποψή μου, έχει ασκήσει πίεση, έχει απλώ την πρόσβαση σε καλά φάρμακα, κυρίω για τα χαμηλότερα στρώματα του πληθυσμού, χαμηλότερα σε οικονομικού πόρου, αλλά τα τελευταία χρόνια η αγορά των φαρμάκων δεν έχει τεράστιες διακυμάνσει. Η αγορά της Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον μια νομοθεσία αποτελεσματική ε, ως προς το θέμα αυτό. Οπότε οι καταναλωτέ, παρόλα αυτά έχουν σοβαρή δυσφορία σε σχέση με την διαθεσιμότητα των φαρμάκων. Ιδίως αυτά που προστατεύονται από δίπλωμα τεχνίας. Έγραψα λοιπόν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκστατεία ευαισθητοποίηση που θα έπρεπε να ξεκινήσει ώστε να, να αποκτήσουν και την απαραίτητη εμπιστοσύνη οι ασθενείς στα απαραίτητα φάρμακα, τα πιο σημαντικά. Και αυτό είναι πραγματικά σημαντικό, ιδίω για όσου δεν έχουν μεγάλη οικονομική άνεση για να προμηθευτούν τα κατάλληλα φάρμακα για τη θεραπεία του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου απήντησε ότι ήδη γίνονται πολλά. Και το ε, επιβεβαιώνουν οι στατιστικέ μελέτε. Ευχαριστώ τη συνάδελφο Καμπεθόν για άλλη μια φορά γιατί καλύπτει όλα τα σκέλη αυτού του πολύπλοκου θέματος και ελπίζω κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει διεξοδικότερα σε όλο το Κοινοβούλιο μια απόμβαση, με μια απόφαση παρέμβασης λίγο πιο δυναμική. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα θέλαμε ευκαιρία να ευχαριστήσουμε και πάλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πολύ σημαντική συμβολή του στο θέμα της πρόσβασης, βελτίωσης πρόσβασης στα φάρμακα. Πολύ αξιόλογο το έργο που έχει γίνει και μεγάλη ενέργεια αφιερώθηκε στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης πρωτοβουλίας. Διαπιστώνουμε επίσης ε, ένα μεγάλο αριθμό τροπολογιών, κάτι που δείχνει την πολιτική ευαισθησία αυτού του θέματος και τις προκλήσεις ε, που θα πρέπει να υπερβούμε προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία. Για το τι πρέπει να γίνει ε, και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα παρατηρούμε ε, μεγάλη σύγκληση ως προς τους στόχους που είναι κυρίως η έγκαιρη πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα για όλους τους ασθενείς και μάλιστα σε δίκαιες τιμές προσιτές διαφυλάσσοντας όμω και την ανταγωνιστικότητα ταυτόχρονα της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας. Όπως, αναφέρεται, όπως αναφέρθηκε και στις 12 Οκτωβρίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και σύμφωνα και με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του περασμένου Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να αναλάβει δράση σε κέριους τομείς που ενδιαφέρουν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα επισημάνω ορισμένου από αυτούς. Καταρχήν, βέλτιστη χρήση ε, της ισχύουσας νομοθεσίας και των αριθμιστικών ε, μηχανισμών για τη βελτίωση για τον ασθενών, της πρόσβασης των ασθενών στα φάρμακα. Επίσης, πρόθεση της καινοτομίας, ε, ιδιαίτερα σε περίπτωση που δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη οι ιατρικές ανάγκες και οι υγειονομικές ανάγκες. Επίσης, η αδειοδότηση για τη θέση εμπορία θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές ε, αποτελεσματικότητας, ε, ποιότητας και διαφάνειας που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε καλή ε, αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων φορέων της αλυσίδας παραγωγής φαρμάκων. Από την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, αδειοδότηση για τη θέση εμπορία και διαδικασίες προσδιορισμού τιμής, επιστροφής, καθώς και φαρμάκο επαγρύπνησης θα πρέπει να αποφύγουμε περιττές ε, επικαλύψεις και έλλειψη συντονισμού, κάτι που καθυστερεί την πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα. Και επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε το περιττό κόστος για τα συστήματα υγείας ε, και τους ε, ερευνητές. Θέλουμε και έχουμε ξεκινήσει μελέτες για, για τα πιστοποιητικά επικουρικής προστασίας και για την ε, διαθεσιμότητα και τις προσιτές τιμές των φαρμάκων. Και μάλιστα θα υποβάλουμε στο Συμβούλιο σήμερα τις μεθοδολογίες ε, και τα χρονοδιαγράμματα των σχετικών μελετών. Φυσικά θα σας κρατάμε ενήμερους για τα πορίσματα αυτών των μελετών. Τέλος, έχουμε και την πρωτοβουλία για την αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας και ε, συμφωνούμε με τον προσανατολισμό και σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη ε, που θα προέλθει από, αυτό, από αυτή σας την έκθεση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη βέβαια και τις ε, διεθνείς μας δεσμεύσεις σε θέματα υγείας και πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά τη γνώμη μας, καλό θα ήταν να γίνει μνήα αυτών των διεθνώς ανηλυμένων υποχρεώσεων και στην έκθεση. Βέβαια δεν είναι εξαντλητικός αυτός ο κατάλογος, αλλά περιμένουμε τις συμβαστικές τροπολογίες ε, για να λάβουμε πιο συγκεκριμένη θέση. Πάντως θα παρακολουθούμε εκ του σύναγκης την όλη διαδικασία και θα αναθεωρήσουμε τη, θέση μας ε, μετά την έγκριση της έκθεσης στην Ολομέλεια. Αν πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, χρήσιμη εμπειρογνωμοσύνη να σας προσφέρει, Είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα στην κυρία Καμπεθόν Ρουίθ ο λόγος. Για άλλη μια φορά. Θα ήθελα να ξεκινήσω και να ολοκληρώσουμε το ίδιο θέμα Τις ευχαριστήσεις προς τους κοιόδης ηγητές για την ε, αμέριστη συνεργασία τους, την αγαστή συνεργασία μάλλον και την ανάγκη που προέκυψε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ε, υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, δεν έχουμε συμφωνήσει σε όλα τα θέματα. Συνεχίζουμε τις συζητήσεις. Για παράδειγμα την πρόταση του κυρίου Πεντιτσίνη για την εξάλληψη της υπατήτητας γάμα ή την πρόθεση κάποιων φαρμάκων που σώζουν ζωές σε πολλές ε, νόσους. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε την ε, εφαρμογή της ιατικής οδηγίας ε, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στα φάρμακα. Έχουμε πολύ έργο μπροστά μας, γιατί 617 τροπολογίες δεν είναι και λίγες, προϋποθέτουν ώρες επεξεργασίας. Πάντως εξακολουθώ να διατρανώνω την καλή μου θέληση για να επιτύχουμε συμφωνία. Γιατί αν θέλουμε ηχηρό και ξεκάθαρο μήνυμα θα πρέπει και η έκθεσή μας να είναι συνεπής. Κάτι που είναι δύσκολο με 617 τροπολογίες από πολλές πολιτικές ομάδες με ε, συμφέροντα που χρήζουν εξισορρόπησης και στάθμισης. Πάντως είναι σημαντικό το τελικό αποτέλεσμα να είναι χρήσιμο, ρεαλιστικό και να δίνει απάντηση Στι προσδοκίες των Ευρωπαϊκών πολιτών, που είναι μια ξεκάθαρη απάντηση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της πρόσβασης στα φάρμακα. Και γι' αυτό είναι απαραίτητη η συνοχή, η συνεργασία μεταξύ μας ε, και αυτό θα επιδιώξω και στις περαιτέρω συνομιλίες. Σας ευχαριστώ. Να σας θυμίσω το φωνοδιάγραμμα. 31 Ιανουαρίου στην ΕΝΒΗ και τον Φεβρουάριο ε, στην Ολομέλεια, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πότε. Πάμε στα διάφορα. Επόμενη έκτακτη συνεδρίαση στις 15 Δεκεμβρίου την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο για να ψηφίσουμε την ε, ε, μεταρρύθμιση του ETS και μετά 12 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες. Μπορούμε να κλείσουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση αλλά εδώ στις 12 σας περιμένω για το χριστουγεννιάτικο κοκτέιλ μας. Ευχαριστώ.